27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 54. Λήξη. Εγκρίνεται. 55. Όχι. Καταπίπτει. 57. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ένας υπεράριθμος στο ΕΛΚ. Εντάξει. Λήξη. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για ηλεκτρονικά για ένα κείμενο συμβασμό συνεισφορά τη ΣΥΤΡΕ στο σχέδιο πρόταση ψηφίσματο τη ΕΝΒΗ, διάσκεψη των Ηνωμένων για την Κλιματική Αλλαγή 2019 στο Σαντιάγο τη Χιλή. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, έρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ και ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Um, I think I will, if we have the next guest... Αν έχει έρθει ο επόμενος ομιλητής, μετά από ένα δύο λεπτά για να αποχωρήσετε όσοι θέλετε για καφέ. Θα περάσουμε. Να με κατευθείαν στο επόμενο θέμα για να έχουμε χρόνο για την συζήτηση και να τελειώσουμε όσο και πιο νωρίς σήμερα. Οπότε ξεκινάμε στο επόμενο θέμα. Okay, thank you very much, colleagues, for taking your seats. Thank you. So we move on with the next item on our agenda, which is a presentation of the Policy Department. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερής διάταξης, που είναι η παρουσίαση μιας μελέτης από το Τμήμα Πολιτικής με θέμα την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε μια βιομηχανική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στραμμένη προς το μέλλον. Η δόκτωρα Τζούλη Πελεγκράν θα μας κάνει τη σχετική παρουσίαση. Ε, εκπώνησε αυτή τη μελέτη μαζί με το Τμήμα Πολιτικής κατόπιν δικής μας αιτήσεως. Η κυρία Πελεγκράν είναι ερευνήτρια στο κέντρο βιομηχανικών σπουδών στο Μιλάνο και έχει διδακτορικό στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και ειδικεύεται σε ανάλυση δημοσίων πολιτικών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας και συντώνησε πολλές εκθέσεις ε, και μελέτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις, επιτροπές Ήτρε και Ρέγγι και μία μελέτη για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική. Η συγκεκριμένη μελέτη που θα μας παρουσιάσει σήμερα ζητήθηκε από τους συντονιστές της Επιτροπής Ήτρε πέρυσι και έχει στόχο την αξιολόγηση της ανακοίνωσης του 2017 που θέμα έχει τις επενδύσεις σε έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία και βιομηχανική πολιτική στραμμένη προς το μέλλον. Μετά την παρουσία της μελέτης θα ακολουθήσει συζήτηση με τη δόκτωρα Πελεγκρά. Κυρία Πελεγκρά, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση για τα ευρήματά μας για το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε προκλήσεις σε μια βιομηχανική στρατηγική για το μέλλον στόχος της ε, μελέτης ήταν να καθοριστεί το εύρος ε, και το περιεχόμενο μιας πολιτικής, μιας βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή καθορίστηκε στην τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2017. Ο στόχος είναι να αξιολογήσουμε το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί η πολιτική αυτή στις μελλοντικές προκλήσεις. Οπότε, θα κάνω το εξής. Ε, θα σας ε, εξηγήσω λίγο το πλαίσιο για να αντιληφθείτε την εξέλιξη της βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης. Θα μπω σε κάποιες λεπτομέρειες ε, για τη μορφή και το περιεχόμενο της, πολιτική, της βιομηχανικής πολιτικής. Θα ασχίσω μετά κάποια κριτική και θα κάνω κάποιες προτάσεις για το μέλλον. Να αναφερθώ λίγο στην μεθοδολογία ε, πρόκειτο για έρευνα γραφείου, συνεντεύξεις ε, προσωπικού της ε, Κομισιόν, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Έγιναν διάφορες μελέτες επίσης στο περιφερειακό επίπεδο, περιπτωσιολογία. Λοιπόν, να σας αναφέρω το πλαίσιο, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από χώρα σε χώρα και μέσα στον χρόνο. Τώρα είμαστε σε μία περίοδο σύνθεσης. Ξεπερνάμε όλες ε, τις ε, διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων ε, των πιο κανονιστικών και των πιο φιλελεύθερων. Έχουμε λοιπόν ένα καλό εργαστήριο θα έλεγα μπροστά μας για να δείξουμε ακριβώς την αλλαγή ε, λογικής για την νέα ε, βιομηχανική πολιτική. Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζετε για το γενικότερο πλαίσιο πέρα από τις ε, νοηματικές εξελίξεις έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η βιομηχανική πολιτική και πάλι δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε βρει τις διάφορες ε, προκλήσεις, ε, τεχνολογικές ε, μεγάλες τάσεις, κοινωνικοπολιτικές τάσεις, παγκοσμιοποίηση, γεωπολιτική, δημογραφία και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Μαζί με συγκεκριμένες προκλήσεις, το Brexit και τα λοιπά που αφορούν ειδικά την Ένωση. Όλα αυτά δημιουργούν κινδύνους, παραδείγματος χάρη εδαφική πόλωση αλλά και ευκαιρίες, ε, π.χ. την δημιουργία νέων αγορών. Έχουμε λοιπόν με βάση αυτά δημιουργήσει τέσσερα κριτήρια για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα της βιομηχανικής πολιτικής, ε, κριτήρια τα οποία θα αναφέρω, τα βλέπετε εκεί στα δεξιά. Αξιολογούμε λοιπόν στρατηγική σύμφωνα με τη δυνατότητα να καθορίσει μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους να αναπτύξει ένα πλαίσιο σύνεπες και συντονισμένο, να μπορεί να προσαρμόζεται στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης. Οπότε, ας ε, δούμε λίγο την ανακοίνωση του 2017 της Κομισιόν που λέγεται «Επένδυση σε μια βιομηχανία έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη» μια νέα βιομηχανική πολιτική για τις Ένωσεις. Έχουν ληφθεί εκ τότε διάφορες ε, πρωτοβουλίες να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η ανακοίνωση του 2017 είναι συνέχεια αυτής της ε, διαδικασίας και το αποκορύφωμά της. Οπότε η ανακοίνωση βρίσκει όλα τα διαφορετικά πεδία πολιτικής που θεωρείται ότι συνεισφέρουν στην ε, βιομηχανική πολιτική της Ένωσης και τα βάζει όλα σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Στην ανακοίνωση υπάρχουν έξι πυλώνες ε, που ε, παρουσιάζονται αλλά είναι χρήσιμο να τους ομαδοποιήσουμε και να δούμε δύο θεματικούς πυλώνες. Ο ένας αφορά την ψηφιοποίηση και την οικονομία χαμηλού άνθρακα και τέσσερις πιο θεματικούς πυλώνες, τα τέσσερα Ά, όπως λέμε, εσωτερική αγορά, διεθνοποίηση, επενδύσεις και καινοτομία. Επίσης, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της ανακοίνωσης είναι η έμφαση που αποδίδει στις ε, συνεργασίες ε, των ενδιαφερομένων κρατών μελών, περιφερειών, πόλεων και της βιομηχανίας βεβαίως. Κοιτώντας τώρα τις ε, διαφορετικές πολιτικές που αναφέρονται εδώ πέρα, βλέπουμε ότι μπορούν να καταταχθούν σε τρεις ε, κατηγορίες δέσμες, αν θέλετε, πολιτικής, που έχουν μια ξεχωριστή λογική, στόχους και παράδοση. Βλέπετε πάνω πάνω στην διαφάνεια πρώτα απ' όλα υπάρχει. Υπάρχουν μέτρα τα οποία ακολουθούν μια οριζόντια προσέγγιση, αφορούν το πλαίσιο, τις συνθήκες κάτι το οποίο καλύπτει και ρυθμιστικά μέτρα αλλά και τις ε, ευρύτερε συνθήκες ε, που αφορούν δεξιότητες, ανθρώπινο κεφάλαιο κτλ. Μια, νέα, μια δεύτερη δέσμη ομαδοποιείται υπό τον τίτλο θεματική και κλαδική προσέγγιση. Εδώ πέρα έχουμε τις παραδοσιακές κλαδικές πολιτικές, π.χ. διαστημική πολιτική, αλλά και μέτρα που έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή που έχουν στόχο να δουν ακριβώς ε, τις ε, κοινωνικές αλλαγές, ε, ψηφιοποίηση, την οικονομία χαμηλού ανθρακά και υπάρχει τέλος και εδαφική προσέγγιση που υπάρχει παρά το ότι δεν τονίζεται πάρα πολύ στην ανακοίνωση όπου βεβαίως ε, λαμβάνουμε υπόψη την εφαρμογή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης ε, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κτλ. Συνολικά λοιπόν αυτά μας ε, δείχνουν μια φιλοδοξία για να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση σε μια βιομηχανική πολιτική με φιλοδοξία να καλύψουμε ένα τεράστιο φάσμα υφιστάμενων πολιτικών. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο συνεκτική και είναι αυτές οι δέσμες, αν υπάρχουν αντικρουόμενοι στόχοι, παραδείγματος χάρη μεταξύ ανταγωνιστικότητας και εδαφικής συνοχής ή και κοινωνικής συνοχής, μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Αυτά είναι παραδείγματα ε, αντιφατικών στόχων που βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, ε, στη διαφάνεια αυτή έχουμε μια ελαφρώς διαφορετική παρουσίαση των ίδιων πολιτικών που παρουσιάζονται εδώ, αλλά τονίζει αυτό κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Κυρίως το ότι κάποιες εξελίξεις ε, στην ε, πολιτική ε, λαμβάνουν χώρα ακριβώς εκεί όπου διασταυρώνονται αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Και έτσι θα έλεγα υπάρχει μια συμφιλίωση των διαφορετικών αυτών αρχών. Οπότε έχουμε μια προσέγγιση της αλυσίδας αξίας την οποία προωθεί η Κομισιόν, δηλαδή εκεί όπου διασταυρώνεται η θεματική και κλαδική προσέγγιση και η προσέγγιση που αφορά το πλαίσιο των συνθήκων. Δηλαδή εδώ πέρα απευθυνόμαστε σε οικοσυστήματα, σε ολόκληρο το μήκος της ε, αλυσίδας ε, παραγωγής από την πρώτη ύλη στο τελικό προϊόν. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις γιατί η αλυσίδα αυτή βεβαίως εκτείνεται σε διαφορετικές χώρες και περιοχές, αφορά διαφορετικούς τομείς πολιτικής και συμμετέχοντες ε, και στο επίπεδο βεβαίως, το εθνικό και το ευρωπαϊκό και το περιφερειακό. Στην διαφάνεια αυτή έχετε μία ένδειξη του προϋπολογισμού που υπάρχει για να στηριχτούν οι διάφορες πολιτικές και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανακοίνωση και βλέπετε την τεράστια σημασία της πολιτικής συνοχής ε, στην χρηματοδότηση. Εντάξει, είναι μια εκτίμηση, αλλά εκτιμούμε ότι ο προϋπολογισμός ο διαθέσιμος είναι γύρω στα 455 δισεκατομμύρια στην περίοδο 2014-2020, τα δύο τρίτα από αυτά είναι από την πολιτική συνοχή. Οπότε βασικά υπάρχει ένα μέσο που ε, προσπαθεί να επιτυχεί τρεις ε, στόχους ε, που ακολουθούν διαφορετική λογική. Αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, με δεδομένα όλα αυτά τα μέτρα και τις πολιτικές και τον ανάλογο προπολογισμό, Ποια διοικητική δομή έχουμε. Η διαφάνεια αυτή μας ε, δείχνει την πρόταση του 2018 που υπέβαλε η Προεδρία. Ενδιαφέρον είναι ότι εμφανίζονται εδώ πέρα νέοι δρόντες, ε, αλλά και ε, τις ημέρες βιομηχανίας ή τη στρογγυλή τράπεζα της βιομηχανίας 2030 που περιλαμβάνει εκπροσώπηση των περιφερειών, των κοινωνικών εταίρων κτλ. και νέε λειτουργίε. Παραδείγματο χάρη, ένα δομημένο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων, η παρακολούθηση με βάση έναν πίνακα βαθμολογίας ε, που περιλαμβάνει πάρα πολλούς δείκτες όλα αυτά είναι προσωρινά και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον λειτουργούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο χρόνος ζωής αυτών των διευθετήσεων περιορίζεται ε, και φτάνει μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Κομισιόν. Οπότε, είτε θα παραταθεί, είτε θα αλλάξει. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο και δεν φαίνεται σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια είναι ότι υπάρχουν πολύ αποκεντρωμένοι μηχανισμοί διοίκησης πλατφόρμες δηλαδή οι οποίες ενώνουν ενδιαφερομένους διαφόρων τύπων ε, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε διάφορα επίπεδα. Παραδείγματο χάρη το στρατηγικό φόρουμ για σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος ε, στη βάση των εξελίξεων αυτών που ανέφερα είναι ένα παράδειγμα. Προσπαθούμε στην έκθεση να έχουμε έναν πλήρη κατάλογο των μηχανισμών αυτών στη σελίδα 64. Οπότε. Συνολικά. Βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες προτεραιότητες ε, που αφορούν κάποιες αποστολές ε, παραγματος χάρη ε, η πράσινη ανάπτυξη κτλ αλλά δεν υπάρχει ακόμα μια επικέντρωση των ε, πόρων και δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος ε, προγραμματισμός που να περιλαμβάνει στόχους ε, και ρεαλιστικούς στόχους. Επίσης η βιομηχανική πολιτική είναι μια μεταπολιτική που αφορά εξτάμενες πολιτικές ήδη. Αλλά είναι ακόμα κάτι το διασπαρμένο και αν υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια συνοχής, όπως μας λέει παραδείγματος χάρη η προσέγγιση αυτή περί της αλυσίδας ε, παραγωγής. Βεβαίως οι εδαφικές ε, πτυχές ε, παραμελούνται. Και τέλος, Βλέπουμε διάφορους αποκεντρωμένους μηχανισμούς που συνεισφέρουν στο να σπάσει η απομόνωση, αλλά αυτό το οποίο λείπει είναι μια γενικότερη ε, διοίκηση και επίσης συντονισμός μεταξύ των περιφερειών. Τέλος, κάποιες σκέψεις για το μέλλον θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνουν ε, κάποιες σοβαρότερες στρατηγικές επιλογές. Υπάρχει μία ανάγκη για έναν ενιαίο στόχο που θα αφορά την κλιματική αλλαγή, καθώς εκεί πέρα είναι το κατεπήγον και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την νομιμοποίηση και την προστιθέμενη αξία. Αυτό πηγαίνει επίσης με ένα ε, σύστημα ε, διακυβέρνησης πιο κεντρικό που θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Το δεύτερο το οποίο θα θέλαμε είναι ότι το περιφερειακό επίπεδο είναι σημαντικό. Εκεί πέρα ε, γίνονται οι ασύμμετροι κραδασμοί, υπάρχουν οι συνέπειες για την κοινωνία και βεβαίω αυτό σημαίνει να δοθεί έμφαση στην στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και τέλος όλα αυτά απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο ε, πολιτικής ε, για να αντιμετωπιστούν ε, οι προκλήσεις που αναδεικνύονται γρήγορα και να προωθηθεί ο πειραματισμός. Σας ευχαριστούμε κυρία Πελεγκρά. Πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη που μας παρουσιάσατε. Και σίγουρα θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση και θα προκαλέσει ερωτήσεις. Κύριε Καρβάλιο ζήτησε πρώτο λόγο. Εδώ δεν μιλώ ως αναπληρώτρια συντονίστρια, αλλά ως απλό μέλος Επιτροπής Ήτρε. Δεν ξέρω αν ε, θέλει ο κύριος Έλλερ πρώτα το λόγο που είναι και συντονιστής. Θέλετε κύριε Έλλερ το λόγο, εγώ διαβάζω το κατάλογο με τους ομιλητές που συνέταξε η γραμματεία. Έχω μια ερώτηση για τη μεθοδολογία της μελέτης αυτής. Μιλήστε για κάποιες ε, συνεντεύξεις που κάνατε σε ό,τι αφορά τους ενεχόμενους, πιθανοί ενδιαφερόμενοι γενικώ ε, από την άποψη δηλαδή της βιομηχανικής πολιτικής ήταν ε, οι συνομιλητές σας ή συμμετείχα σε μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική γιατί αλλάζει έτσι το πρίσμα της ε, μελέτης ανάλογα με το φάσμα των ενεχομένων που εξετάσατε, αλλάζει και η σκοπιά της μελέτης. Ποιοι, ποιοι ήταν οι συνομιλητές σας. Ήταν συγκεκριμένοι βιομηχανικοί τομείς ή ενεχόμενοι ε, κάποια συγκεκριμένη βιομηχανικής πολιτικής. Μας ενδιαφέρει με ποιους ήρθατε σε επαφές. Γιατί είναι δυνητική δικαιούχοι ε, οι ενεχόμενοι που αναφέρεται, οι ενδιαφερόμενοι ή ήδη συμμετείχαν σε ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και ήταν ε, επωφελούμενοι από την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική ήδη. Επίσης, ό,τι αφορά τη μόχλευση και τη διακυβέρνηση, Ποια ήταν τα πόρισματά σας σε ό,τι αφορά την αυτοδιοργάνωση, τη διαδικασία διακυβέρνηση στην Επιτροπή. Και έχω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα έχουμε μιλήσει για μια πολιτική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στη βιομηχανία και υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί, μέσα και χρηματοδότηση για το χάλιβα. Ε, για χαλιβοργίες που δεν θα παράγουν διοξίδιο του άνθρακα, αλλά τέσσερις γενικοί διευθυντές δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε, στη χρηματοδότηση, ώστε όντως ε, να εγκριθεί ένα σχέδιο για χαλιβουργία χωρίς διοξίδιο του άνθρακα, που ήταν αναγγελθεί στόχος της βιομηχανικής πολιτικής. Ποια ήταν τα διδάγματά σας, αντιλήσατε κάποια διδάγματα από την ε, διαδικασία εσωτερικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι υπάρχοντες μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς ή όχι. Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε μια αξιολόγηση ε, για να αντιληφθούμε και πόσο συνεκτική ήταν η μελέτη σας. Ευχαριστώ κύριε Τόγια. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Όπως και η πρόεδρος Βαλεάν, θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη αυτή που μας κάνει να σκεφτούμε τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι ως Ευρώπη και τι δεν έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική στρατηγική γιατί σίγουρα μεταξύ των ε, τομεακών πολιτικών ε, ή των, ε, του γενικού χαρακτήρα εργαλείων που αφορούν τη βιομηχανία, εμείς αυτά τα χρόνια δεν έχουμε ένα στρατηγικό όραμα δηλαδή ολοκληρωμένα μέσα και ολοκληρωμένους στόχους, ολοκληρωμένο όρημα. Θέλω να αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία. καταρχήν, εσείς είπατε ότι έλειπε η εξή πτυχή, μία ολοκλήρωση των μέσων που είναι απαραίτητα για τη βιομηχανική πολιτική και τη εδαφική συνοχή. Είπατε τα δύο τρίτα είναι εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης, φαντάζομαι ότι το άλλο τρίτο είναι έρευνα και καινοτομία, όμως εμείς δεν τα έχουμε ολοκληρώσει αυτά. Αυτό είναι ένα δύναμο σημείο, πώς να το κάνουμε. Όμως αντίθετα μεταξύ των οικονομικών και βιομηχανικών πολιτικών και της κοινωνικής συνοχής υπήρξε κάποια αναφορά. Γιατί τώρα εμεί θα εργαστούμε πολύ στο θέμα αυτό. Παραδείγματο χάρη, σκέφτομαι και την κοινωνική συνοχή για τι περιβαλλοντικέ πτυχέ. Μιλάμε ήδη για διάφορα τέτοια θέματα, δηλαδή πώ θα γίνει αυτό ο συσχετισμό και πώς θα, να δούμε πώς θα συνδέσουμε καλύτερα στόχους βιομηχανικής πολιτικής ε, και κοινωνικής συνοχή. Και το τελευταίο σημείο αφορά τις στρατηγικές πτυχές. Είπατε ότι ε, οι επιλογές ε, για την κυκλική οικονομία και η συμμαχία για τις μπαταρίες ήταν αδύναμα σημεία. Εμείς ε, θέλουμε να ενδυναμώσουμε καταρχήν την ευρωπαϊκή βιομηχανία πριν να έρθουν να μας κατακτήσουν οι Κινέζοι όπως έγινε με τα ηλιακά πάνελ στην ε, μελέτη σας ε, ποιους άλλους κλάδους θεωρείτε ότι θα χρειάζεται μια μεγάλη συμμαχία από τον ε, παραγωγικό κόσμο έτσι ώστε να προωθεθεί η βιομηχανία στην Ευρώπη. Αυτό θα μας ενδιαφέρει. Επίσης συγχαρητήρια να σας πω γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμη η μελέτη αυτή για τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ κυρία Τόγια και κυρία Νταμπάλοβα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Πελαγκράν για την παρουσίαση της μελέτης ενδιαφέρουσα πολύ. Έχω κάνα δύο ερωτήσεις. Μάλλον θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο στη συζήτηση γιατί είναι περισσότερο φιλοσοφικού χαρακτήρα. Αλλά θα ήθελα να μάθω. Μας λείπει μια συνέργεια μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και μηχανισμών. Πού έγκυται το βασικό πρόβλημα, η αδυναμία στη συνέργεια. Στα εδάφη, στις περιφέρειες, ε, στα ερευνητικά προγράμματα σχέση με τη συνοχή πολιτική. Πού υπάρχουν τα χάσματα της συνέργειας, πού τα εντοπίσατε εσείς. Δεύτερον, πώς ε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε επαρκή κάλυψη και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανική πολιτική και στις κατευθυντήριες γραμμές που δίνουμε. Γιατί, ναι, μεν μιλούμε για τη βιομηχανία, αλλά μην ξεχνούμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα μεριμνήσουμε και θα εξασφαλίσουμε και δική τους κάλυψη. Ε, υπάρχουν πορίσματα για μια διαφορετική προσέγγιση ε, της βιομηχανικής στρατηγικής από πλευρά των κρατών μελών. Φαντάζομαι, ναι, θα είναι διαφορετική προσέγγιση των κρατών μελών, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα πορίσματα για το πού έγινε αυτές οι διαφορές. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορέ μεταξύ παλιών και νέων χωρών μελών σε ό,τι αφορά την βιομηχανική στρατηγική του, γιατί έχουν διαφορετική βιομηχανική βάση, οπότε φαντάζομαι υπάρχουν διαφορέ. Αλλά διερευνήσατε τι διαφορέ αυτέ περαιτέρω. Και τέλο, πώς θα εμπλέξουμε καλύτερα στη συζήτηση τη βιομηχανία και τους ενδιαφερόμενους, τους ενεχόμενους. Είναι επαρκής οι προσπάθειές μας. Γιατί οι ενεχόμενοι δεν ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τους ηθήνοντες πολιτικής ή οι ηθήνοντες πολιτικής κοφεύουν στα αιτήματα των ενεχομένων. Πώς θα εξασφαλίσουμε καλύτερη επαφή μεταξύ τους, ώστε να έχουμε περισσότερο feedback και προτάσεις από την ίδια τη βιομηχανία, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους δηλαδή. Ευχαριστώ. Κύριο Νινίστο προηγείται μια συνάδελφος, η κυρία Χάν. Καλώς, η κυρία Χάν τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θαυμάσια αυτή παρουσίαση. Για εμένα είναι σαφές, ε, χρειαζόμαστε μια στρατηγική η οποία θα είναι οικολογική και κοινωνική παρουσίαση μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και πραγματικά μας δείχνει το τι είναι δυνατόν, πού υπάρχουν οι δυνατότητες. Βεβαίως εμένα με ενδιαφέρει αν έχετε την δυνατότητα να κάνετε τρεις προτάσεις. Πώς θα δημιουργήσουμε συνέργειες, συμμαχίες, πώς ε, θα προωθήσουμε την προστασία του κλίματος και τι κοινωνικής προδιαγραφέ. Με συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορείτε να μας πείτε εδώ πέρα μπορούμε να προωθήσουμε κάτι ως πολιτική. Και τι μπορεί να γίνει ως μέτρο για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ. κύριο Στοσενόφσκι, είδα ότι ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Στομπισόφσκι θα μιλήσει εκ μέρους των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για την παρουσίαση, κυρία Πελεγκράν. Νομίζω ότι πολύ σημαντική είναι αυτή η βιομηχανική στρατηγική και θα πρέπει να κάνει μια διάγνωση των ε, προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Θα πρέπει να γίνει καλύτερη συνα... Ε, καλύτερος συνδυασμός μεταξύ της πολιτικής στήριξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, είχαμε την στρατηγική 2025 της Κίνας για την μεταποιητική της βιομηχανία ή την προστατευτική πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ε, ε, οικονομίες και απόψη καινοτομία. Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία επίσης είναι σημαντικοί ανταγωνιστές. Οπότε στις εμπορικές μας συμφωνίες θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη και να στηρίξουμε και τη δική μας βιομηχανία. Ε, Μήπως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σκεφτεί πιο αναλυτικά αυτά τα παραδείγματα των ανταγωνιστών της και να λάβει υπόψη και να εκπονήσει το δικό της χαρακτηριστικό μοντέλο της βιομηχανίας της. Γιατί για τα πολλά τελευταία χρόνια δεν είχαμε νέες επιχειρήσεις σε καινοτόμους ανταγωνιστικούς τομείς. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δικό μας μοντέλο εξάπλωσης της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πιθανότητες βλέπετε για να αλλάξει μέχρι τώρα κατάσταση. Κατά τη γνώμη σας, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τους δικούς μας πρωταγωνιστές από τους, τους ευρωπαϊκούς, δηλαδή από τους άλλους εθνικούς πρωταγωνιστές. Επίσης, πώς θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη κάποιων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θα είναι πρωταγωνιστές και πρωτοπόροι. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος. Περνάμε στο δεύτερο γύρο. Σε λίγο θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Πελεγκράν για να απαντήσει στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων και μετά θα έχουμε και δεύτερο γύρο. Καταρχήν, δύο λόγια για τη μεθοδολογία. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις με τη σειρά που τέθηκαν. Είναι μια σχετικά μικρή μελέτη. Δεν είχαμε ούτε το χρόνο ούτε τα μέσα ε, για να έχουμε πραγματικά αντιπροσωπευτικές ε, διαβουλεύσεις με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων ενεχομένων. Αυτό που προσπαθήσαμε είναι να επικεντρωθούμε σε, εθνικό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τους ε, ε, και σε εθνικό επίπεδο ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους κάποιων ε, ε, ομοσπονδιακών οργάνων ε, βιομηχανικών. Και επίσης ήρθαμε σε επαφή με κάποιους εκπροσώπους περιφερειακών βιομηχανικών κλάδων για να δούμε πόσο σημαντικό είναι το θεσμικό περιβάλλον και πώς επηρεάζει τα διάφορα μέτρα ή πώς αξιοποιεί τα διάφορα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ε, το θεσμικό υπόβαθρο των μέτρων είναι πολύ σημαντικό και το πώς εντάσσεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες. Και αυτό είναι ο γνώμονα τη αποτελεσματικότητα ενός μέτρου. Μπορεί να έχει κανείς κατάλληλα μέτρα πολιτικής, αλλά θα πρέπει να είναι αυτά κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες, στις περιφερειακές ανάγκες, στις τοπικές ανάγκες και να γίνονται και δεκτά εκεί και να είναι πρόσφορο το θεσμικό περιβάλλον για να διευκολύνει αυτή την αποδοχή και τη σωστή εφαρμογή. Η εσωτερική διαδικασία διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπατε ποια είναι. Έγιναν κάποιες διαβουλεύσεις, ε, συνεντεύξω αν θέλετε, με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τις επαφές αυτές διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια πρόοδος ε, και μεγαλύτερη συνεργασία πια μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί όντως το παρελθόν, σε μια προηγούμενη μελέτη που είχαμε εκπονήσει για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική, είχαμε τότε διαπιστώσει πριν από μερικά χρόνια ότι δεν ήταν εμφανή η συνεργασία μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων. Υπήρχε μια στεγανοποίηση. Τώρα υπάρχει πολύ καλύτερη επικοινωνία και καλύτερο συντονισμός μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Δεν υπάρχουν βέβαια κάποιοι επίσημοι μηχανισμοί, τυπικοί μηχανισμοί. Είναι όλα άτυπα όλες αυτές οι επαφές και ο συντονισμός γίνεται άτυπα, δεν είναι θεσμοθετημένα. Αλλά υπάρχουν τέτοιε επαφέ μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάγκη συνδυασμού και συμφιλίωσης της κοινωνικής συνοχής με τη βιομηχανική πολιτική. Για να είμαι ειλικρινής, το πόρισμά μας κρίνει αυτό το σημείο ως αδυναμία της τρέχουσας στρατηγικής και φαίνεται και στην ανακοίνωση του 2017. Και αν κανείς προσπαθεί ε, βάλει την, τον όρο συνοχή για την, στην αναζήτηση στο ίντερνετ, δεν θα βρει και πολλές μνήες. Η εδαφική συνοχή, αμελείται, αλλά δυστυχώς παραμερίζεται, παραγωνίζεται και η κοινωνική συνοχή στη βιομηχανική πολιτική. Οπότε αυτή την ε, απόσταση θα πρέπει να την διορθώσουμε. Και είναι πολύ σημαντική η πολιτική συνοχής από άποψη χρηματοδότησης, αλλά η πολιτική συνοχή είναι κυρίως, έχει κυρίως εδαφική διάσταση, όχι τομεακή Οπότε η μόνη διάσταση που είναι πραγματικά εδαφική και αναφέρεται στην ανακοίνωση του 2017 είναι οι στρατηγικές έξυπνης ειδίκευση. Τώρα, που υπάρχει χάσμα συνεργειών, που είναι οι βασικές αδυναμίες. Εμείς έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερως με την πολιτική συνοχής και εξετάζοντας την κατάσταση σε περιφερειακό επίπεδο, είναι φανερό ότι είναι δύσκολο να συνδυαστούν τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που υπάρχουν. Από την πολιτική συνοχής, από τον ορίζοντα 2020. Είναι διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμοί με διαφορετικούς σκοπούς και δεν υπάρχει καλό συνδυασμό μεταξύ του. Δεν υπάρχει ολοκλήρωση, δεν υπάρχει συνδυασμό ούτε σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει ελάχιστο ή μερικές φορές και μηδενικό συντονισμό μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε εκεί υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στη συνέργεια και υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Γι' αυτό και είπαμε ότι υπάρχει η ανάγκη σωστής δομής και διακυβέρνησης για το συντονισμό των διάφορων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όντως ε, δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θεωρητικά καλύπτονται από την πολιτική συνοχής και μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ορίζοντα 2020. Και έχουμε και τη χρηματοδότηση από τον οργανισμό ΕΑΣΜΕ, που είναι ειδικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Τώρα, ε, διαφορετικές προσεγγίσεις από τα κράτη-μέλη και συγκεκριμένες διαφορές. Μιλήσαμε για την ανάγκη να προωθήσουμε και να δείξουμε Ευρωπαίους πρωταθλητές, Ευρωπαίους πρωτοπόρους, πρωταγωνιστές. Η γαλλική προσέγγιση είναι το γαλλικό σήμα εμπιστοσύνη που δίνει ενάυσματα για πρωτοπόρες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω γνωρίζετε μια γαλλογερμανική διαμαρτυρία κατά της απόφασης να μην επιτραπεί μια μεγάλη συγχώνευση για να δημιουργηθεί ένας τέτοιος Ευρωπαίος πρωταθλητής. αυτό είναι ένα παράδειγμα διαφορετικών προσεγγίσεων στη βιομηχανική πολιτική. Άλλη προσέγγιση θα ήταν ε, λήψη υπόψη περιφερειακών κριτηρίων ή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα, πώς θα εμπλέξουμε καλύτερα τους ενδιαφερόμενους, τους stakeholders. πολλά γίνονται μέσω του κεντρικού μηχανισμού και πολλά θα πρέπει να γίνουν και περισσότερα σε υψηλότερο επίπεδο. Είναι θέμα διακυβέρνησης δηλαδή. Τρία πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν, που θα έπρεπε να αλλάξουν. Τώρα τρία συγκεκριμένα δεν ξέρω, αλλά όπως προκύπτει και από την παρουσίαση που σας έκανα, το πρώτο που θα πρέπει να αλλάξει είναι να μεριμνήσουμε για να έχουμε μια σωστή στρατηγική διακυβέρνηση, η μορφή διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό θα αποφασιστεί σχετικά σύντομα. Και εκεί υπάρχει περιθώριο βελτίωση και λιγμών και για σας για να επηρεάσετε την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν κάλυψα όλες τις ερωτήσεις και έχασα τίποτα. Να ακούσουμε και του υπόλοιπου συναδέλφου. Κύριε Καρβάλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση της μελέτης. Έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Ωστόσο, νομίζω ότι κάτι λείπει και έχει να κάνει με την τεχνολογική ηγεσία. Προκειμένου να έχουμε μία βιομηχανική πολιτική, πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε ηγετική θέση στους τομείς που την έχουμε ήδη κατεκτήσει και να ξανακερδίσουμε την ηγετική θέση σε κάποιους τομείς. Αυτό το κάνεις μέσω της έρευνας και τεχνολογίας. Έχουμε παραδείγματα παραδείγματα που είμαστε σε ηγετική θέση, πρέπει το χάρη στην αυτοκίνητο βιομηχανία, υπάρχουν επενδύσεις ε, σε επιδείξεις κτλ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτή την ηγετική θέση λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό λείπει. Η τεχνολογία, ε, νέες τεχνολογίες που πρέπει να αναπτύξουμε για να ανταγωνιστούμε με την ε, Νότιο Κορέα, το χάρη. Το δεύτερο σχόλιο μου είναι ότι έχετε ένα μοντέλο διακυβέρνησης. Αν μιλάτε ε, για τη διακυβέρνηση των κονδυλίων, συμφωνώ. Αν μιλάτε για το μοντέλο που αφορά τη βιομηχανική πολιτική και τη σχετική διακυβέρνηση, δεν συμφωνώ τόσο πολύ. Πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται η βιομηχανία είναι ε, χώρος να αναπνεύσει, να μην έχει εμπόδια στην ανάπτυξη. Φυσικά υπερασπίζουμε και το περιβάλλον ε, και τα κοινωνικά ζητήματα. Δεν θέλουμε να έχουμε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, ε, ούτε τον κεντρικό σχεδιασμό που περιγράψατε. Βλέπω και δύο τομείς που θεωρώ ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Δεν τονίστηκαν ιδιαίτερα στη μελέτη σας να εξετάσουμε το θέμα του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε και το πώς σχετίζονται αυτά με την έρευνα και την ανάπτυξη και να δούμε και το εμπόριο. Και τι γίνεται στο θέμα της αμοιβαιότητας στο εμπόριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουταχάρ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Πελεγκρόν για τη μελέτη και την παρουσίαση. Όντω ε, το να διαμορφώνουμε την ε, βιομηχανική πολιτική και την τεχνολογική βιομηχανία είναι κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο. Το ίδιο ισχύει και για την, ε, το θέμα της κυριαρχίας, αλλά και το να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον θα εργαστεί στο θέμα της τεχνολογικής κυριαρχίας και θα επικεντρωθεί σε κάποιους κρίσιμους τομείς. Μου άρεσαν οι συστάσεις που περιλαμβάνονταν στη μελέτη σας και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο να έχουμε πιο ακριβείς στρατηγικές επιλογές και να συνεχίσουμε τον πειραματισμό. Θεωρώ ότι αυτές οι συστάσεις μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να έχει ένα υγιές τεχνολογικό μέλλον. Και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική, θέλω να σας ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση ποια εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να πετύχει αυτή την τεχνολογική κυριαρχία, πώς μπορούν να συνεισφέρουν ε, όσοι χαραζούν την πολιτική και ποιες ε, είναι οι εθνικές προσπάθειες στον τομέα αυτό. Μιλώ για τη δέσμευση των περιφερειών και των κρατών μελών σε όρους βιομηχανικής πολιτικής. Ποια είναι η συνεισφορά οι γεωγραφικές περιφέρειες, τα νησιά μπορούν να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς μιλάμε και για μια τεχνολογική μεγατάση. Σας ευχαριστώ κυρία Τσέχ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και μου άρεσε που τονίσατε τη σημασία των περιφερειών και των διαρθρωτικών ταμείων. Ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θα ήθελα να ακούσω ποια ήταν τα συγκεκριμένα προβλήματα που θα μπορούσατε να τονίσετε που έλαβαν χώρα ε, στις προηγούμενες θητείες ποια ήταν τα προβλήματα που δεν μπόρεσαν να επιτρέψουν το συντονισμό και τι θα πρέπει να κάνουμε ως νέοι νομοθέτες σε αυτή την θητεία. Συγκεκριμένα, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να διορθωθεί η έλλειψη συνεργειών. Μιλάμε μόνο για περισσότερη επικοινωνία, νέα προγράμματα. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες ε, χώρες να ξεπεράσουν την καθυστέρηση και να δημιουργήσουν πραγματικά ολοκληρωμένη και πιο ισότιμη ε, βιομηχανική πολιτική, βιομηχανικό τοπίο. Ευχαριστώ. Η κυρία Τελκαστήγιο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έρχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή, καθώς ξεκινάμε την εθιτεία. Αφενός αφετέρου, αυτή την εβδομάδα έχουμε και τις εκροάσεις με τους υποψήφιους επιτρόπους. Κατά την άποψή μου, αυτό που είναι πολύ τόσο απαραίτητο και λείπει σε αυτόν τον ε, ωκεανό τη ε, βιομηχανική πολιτική. Μιλάτε για τη βιομηχανική πολιτική και ουσιαστικά όταν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για έναν ωκεανό. Και ο καθένα μα πρέπει να αναρωτηθεί τι γίνεται με την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Έχετε μία τέτοια μελέτη και στην παρουσίαση έπρεπε να τα αναφέρετε αλλά δεν μπορείτε να εξηγήσετε πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική με έναν συνολικό τρόπο. Πρέπει να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα πράγματα, να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τα κύρια χαρακτηριστικά μίας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, γιατί αυτό είναι όρος πολιτική. Εμείς χρειαζόμαστε, κατά την άποψή μου, ένα θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική ακριβώς όπως είχαμε το 2009 με το ψηφιακό θεματολόγιο. Ή με όλες τις συγκεκριμένε προτάσεις για την κλιματική αλλαγή και τις σχετικές δράσεις ή στον ενεργειακό τομέα κτλ. Χρειαζόμαστε κάτι που θα είναι ολοκληρωμένο και θα είναι έτσι προσδιορισμένο έτσι ώστε να μπορούμε να θέτουμε στόχους και τα κατάλληλα μέσα για να φτάσουμε στους στόχους αλλά και την κατάλληλη χρηματοδότηση και αυτό σε βραχυπρόθεσμο, μεσοκρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Και όλοι μας τότε θα έχουμε μία πιο ξεκάθαρη ιδέα για το τι χρειάζεται από το, από θεσμικό όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μπορέσουν να συνεισφέρουν να γίνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Αλλά αυτό χρειαζόμαστε. Αν δεν το έχουμε αυτό, τότε θα βρισκόμαστε συνεχώς στην ίδια κατάσταση. Και δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο ωκεανό. Θα γίνει μάντρα τελικά η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για μας. Αυτή είναι η πρότασή μου, να έχουμε ένα θεματολόγιο λοιπόν. Θα ήθελα τη γνώμη σας επ' αυτού. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έχουμε εδώ, ο κύριος Μπλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Πελεγκρίν. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ερώτηση που έκανε η συνάδελφος. Είπατε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες στρατηγικές επιλογές ε, και αναφερθήκατε σε μια καλύτερη διοικητική δομή. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε τι εννοείτε με αυτό, τι, μορφή θα έχει. Ε, λίγο να το τεκμηριώσετε. Και μετά η άλλη ερώτηση. Αναφερθήκατε σε αυτά τα θέματα όπως το πράσινο New Deal, ε, που είναι βεβαίως ε, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και η μεγαλύτερη ευκαιρία που αφορά ακριβώς την απομάκρυνση από τον άνθρακα. Αν δούμε λοιπόν την τρέχουσα κατάσταση της ε, πολιτικής και την ε, δομή, την διοικητική, είναι αρκετά ευέλικτη αυτή η δομή για να ανταποκριθεί σε τέτοιες προκλήσεις και πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσει να προσαρμοστεί στην βιομηχανική πολιτική άλλων χωρών όπως της Κίνας και λοιπά. Σας ευχαριστώ κύριο Πίπερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις βάσεις ε, με τις οποίες μπορούμε να χαράξουμε την πολιτική μας. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω να σκεφτούμε λίγο περισσότερο από τη, να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τις επιχειρήσεις. Το θέμα είναι η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών στην Ευρώπη που θέλουν να εξάγουν, που θέλουν να δημιουργούν α, ε, θέσεις εργασίας ε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ε, του κλίματος, με την εμπορική πολιτική, με την ψηφιοποίηση, αλλά χρειάζεται μια στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με όλα αυτά τα ζητήματα. Και εκεί πέρα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Δεύτερη και τελευταία παρατήρηση είναι εξής. Ε, κοιτάξτε, πάλι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιορίζονται σε startups, ε, στο Horizon ε, και, τα και στα λεφτά. Όχι. Μια πολιτική για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κάτι παραπάνω. Πρέπει να ασχοληθεί με το δίκαιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την εμπορική πολιτική, με την ρύθμιση. Σε όλους τους ε, τομείς, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε για την προστασία των δεδομένων, δεν υπάρχει μια λογική τέτοια πολιτική πραγματικά θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε αντί να περιοριζόμαστε μόνο στα λεφτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πίπερ. Τώρα η κυρία Σόλις Πέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μελέτη αυτή. Το ερώτημά μου αφορά την εδαφική συνοχή το έθεσαν ήδη οι συνάδελφοι και ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακών Ζητημάτων θα ήθελα ακριβώς να γνωρίζω αυτές τις μεγάλες τάσεις ε, που θα μπορούσαν βεβαίως να επιφέρουν μια, κοινωνικό κατακαιρματισμό. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, αλλά όχι ει βάρο της ε, εδαφικής ε, συνοχής. Η άλλη ερώτηση ακούστηκε ήδη αφορά τις συνέργειες. Τι μπορεί να γίνει για να διευκολύνουμε τι συνέργειες μεταξύ βιομηχανική ε, πολιτικής και της πολιτικής της βιομηχανικής και της έρευνα και ανάπτυξη και για να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που συχνά είναι πάρα πολύ χαμηλή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα και ο Σκουρμπιλίους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ για την μελέτη και για την ε, συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε μια σαφή αντίληψη των μεγάλων ε, προκλήσεων ε, και των στρατηγικών στόχων. Υπάρχουν ακριβώς ε, αυτά τα έγγραφα στρατηγικής του 2017, πολλά πράγματα για την ε, διοίκηση, αλλά λίγα πράγματα για τις σοβαρές ε, προκλήσεις και τους λόγους αυτές. Γι' αυτό το λόγο Εγώ διάβασα πρόσφατα τη γερμανική βιομηχανική στρατηγική που είναι ε, πολύ πιο ξεκάθαρη και θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ πιο προσεκτικά και την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Τι σκέφτεσαι για την ε, σχέση μεταξύ της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανικής πολιτικής και των εθνικών στρατηγικών και πώς θα αποφευχθεί εδώ πέρα μια αντίφαση. Οι Γερμανοί μιλάνε πάρα πολύ για το πώς οι εταιρείε, οι παγκόσμιοι ανταγωνιστικές αντιμετωπίζουν προκλήσεις, πώς θα δημιουργηθούν ε, γερμανικές ε, και ευρωπαϊκές εταιρείε και στην εμπειρία μας μέχρι στιγμής ε, η, η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εναντίον ενός τέτοιου ενδεχομένου. Οπότε υπάρχουν πολύ σοβαρότερα φιλοσοφικά ερωτήματα από την διοίκηση απλώς ε, της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής που δεν έχω καταλάβει ακριβώς ε, τι αφορά. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να δω πώς η γερμανική βιομηχανική πολιτική θα μπορούσε να επεκταθεί και να αποτελέσει μια... Ευχαριστούμε κύριε Κομπίλους. Τελευταίο ομιλητής. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά, κυρία Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει ένα λυσαλαίο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 20% ε, είναι η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό έπανο, στην Κίνα είναι 42%, στη Ρωσία είναι 32%. Εξού και αυτός ο ε, λυσαλαίος και δυσανάλογος ανταγωνισμός ε, σε παγκόσμια κλίμακα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική. Γιατί θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην εξέταση τη ευρωπαϊκή αγορά, γιατί είμαστε τμήμα μια παγκόσμια αγοράς και σε τέτοια κλίμακα παγκόσμια θα πρέπει να βρούμε κάποιε λύσει για τη βιομηχανία μα. Επίση θέλουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ τη εμπορική και τη βιομηχανική πολιτική, ώστε να αποτρέψουμε περαιτέρω μετεγκαταστάσει εργοστασίων και μια αποβιομηχάνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη σας, μια φιλόδοξη βιομηχανική στρατηγική δεν χρήζει μιας μεταρρύθμισης στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου για να εξασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού και σε ό,τι αφορά το άνοιγμα στις δημόσιες συμβάσεις και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Για παράδειγμα, η Κίνα μας εντυπωσιάζει στον τομέα αυτό, γιατί η Κίνα ε, επιτίθεται στο σιδηροδρομικό μας κλάδο και μας πουλάει τρένα. Ενώ είναι κλειστή η αγορά δημοσιοσυμβάσεων ε, στην Κίνα. Οπότε να ελέγξουμε τις κρατικές ενισχύσεις, ε, να προωθήσουμε το ρόλο των δημόσιων επιχειρήσεων και να δούμε και την αναγκαστική μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Ευχαριστώ. Κύριε Πελεγκράμ. Προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες και εύστοχες ερωτήσεις. Νομίζω ότι είναι τόσο απέραντος αυτός ο τομέας που είναι λογικό να επισύρει πολύ άριθμες ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά την ηγετική μας θέση στην τεχνολογία και κάποιους τομείς επιμέρους Δεν ξέρω θα πρέπει να εμείνουμε σε αυτή την έννοια την τομεακή ή αν κρατήσουμε κάποιες τομεακές πολιτικές που είναι αιτιολογημένες, παρόλα αυτά θα πρέπει να τις συμπληρώσουμε με μία νέα ενιαία ανάλυση και να ξεπεράσουμε τα στενά όρια των τομέων, να έχω μία ευρύτερη ανάλυση διατομεακή. Για παράδειγμα, έχουμε κάποιες νέες τάσεις στα όρια κάποιων τομέων. Έχουμε αναδυόμενες βιομηχανίες που δημιουργούνται συνδυάζοντας κάποιες ειδικότητε, ε, κάποιους τομείς. Δεν είναι στεγανός λοιπόν ο διαχωρισμός των τομέων. Η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική λοιπόν δεν θα πρέπει να στρέφεται σε συγκεκριμένους τομείς αν θέλει να έχει ηγετική θέση παγκοσμίω. Βέβαια δεν θα πρέπει να γίνει μια να εφαρμοστεί ή να επιβληθεί μια κεντρική προσέγγιση από την κορφή προς, προς τα κάτω. Χρειαζόμαστε όμως ένα παγκόσμιο όραμα και ένα θεματολόγιο, όπως είπατε. Και λαμβάνουμε υπόψη το γενικό πλαίσιο και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Δεν είναι ότι θα επιλέξουμε συγκεκριμένους τομείς ή κλάδους ή περιοχές. Και στο θεματολόγιο αυτό υπάρχει, όπως είπατε, περιθώριο και για τις περιφέρειες. Δεν θέλουμε ένα κεντρικό σχεδιασμό, αλλά ένα καλύτερο κεντρικό συντονισμό των των μέσων. Και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εκ του μηδενός μια βιομηχανική ευρωπαϊκή πολιτική. Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική είναι μια μεταπολιτική, δηλαδή στηρίζεται στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και περισσότερο έχει νόημα ένας καλύτερος συντονισμός των ε, ισχυωσών πολιτικών. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κρατικές ενισχύσεις ε, και τον ανταγωνισμό, υπάρχει τρόπος να συμφιλιώσουμε και να συνδυάσουμε αντικρουόμενα συμφέροντα. Για παράδειγμα, ε, σας μίλησα για την, για την προσέγγιση της αλυσίδας αξίας. Αυτό είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε το εμπόδιο των κρατικών ενισχύσεων με κάποιες ειδικέ ρυθμίσεις για, την, για τις εξελίξεις και στον τομέα αυτό. Οι περιφέρειες τώρα. Αυτό που προκύπτει από τη μελέτη μας και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με το θέμα αυτό για το λόγο αυτό ακριβώς γιατί είχα εμπειρία με την περιφερειακή ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής. Και όταν ε, αν επικεντρωθούμε στο τι συμβαίνει μόνο στις περιφέρειες, χάνουμε το συνολικό όραμα των διαφορετικών περιφερειών που προσπαθούν να αναπτυχθούν όπως μπορούν η καθεμία. Αυτό όμως που λείπει είναι καλύτερη διακυβέρνηση του διαπεριφερειακού συντονισμού. Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες, όπως η πλατφόρμα της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκεί έχουν επαφές οι περιφέρειες μεταξύ τους και ή ευθυγραμμίζονται ή αξιοποιούν ε, τις θετικές τους εμπειρίες. Αυτό είναι σημαντικό. Αλοχεύει όμως ο κίνδυνος είναι πολύ κατακαιρματισμένες ε, αυτές οι πρωτοβουλίες και μεμονωμένες και ουσιαστικά κάθε περιφέρεια δουλεύει δηλαδή μόνη της. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν πιο κεντρικό συντονισμό των διαπεριφερειακών σχέσεων και των διαπεριφερειακών πρωτοβουλειών. I can just agree. Συμφωνώ με την ανάγκη να επικεντρωθούμε στις επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και υπάρχουν πολλά μέτρα που δικαιώνουν τις ευρωπαϊκές δράσεις στον τομέα αυτό, αλλά δυστυχώς τα προγράμματα είναι λίγο κατακαιρματισμένα. πώς θα βελτιώσουμε την ικανότητα των περιφερειών να απορροφούν κονδύλια. Πώς θα ενισχυθεί η ικανότητα εκταμείευσης των περιφερειών. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κατάλληλη πολιτική, ε, ικανότητα πολιτικής σε πολλά επίπεδα και σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό. δεν αρκούν μόνο καλά μέτρα πολιτικής ή σωστέ ρυθμίσεις διακυβέρνησης. Θα πρέπει οι ηθήνοντε της πολιτικής να είναι αρκετά δεκτική, να είναι ανοιχτοί και να μπορούν να, να εφαρμόσουν τα μέτρα ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει αυτό που κάνει ήδη η πολιτική συνοχής, την τεχνική αρρωγή. Θα πρέπει οι περιφέρειες να βελτιώνουν την διοικητική τους ικανότητα και να μαθαίνουν συνεχώς, όχι μόνο σε περιφερειακό μας επίπεδο. τι μια ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική, ρωτήσατε. Δεν αρκούν εθνικές βιομηχανικές στρατηγικές που φαίνονται απλούστερες και πιο συγκροτημένες. Υπάρχει προστιθέμενη αξία σε μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. η ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να επιφέρει προστιθέμενη αξία και η προστιθέμενη της αξία έγκυται ακριβώς στην ανάδειξη της ισχύω των περιφερειών και των χωρών. Αλυσίδες αξίας, για παράδειγμα, που είναι διακρατικές. Είναι καλό παράδειγμα αυτής της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Επίσης θα μπορούσαμε να βρούμε λύσεις για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές για να κερδίσουν το χαμένο έδαφος και να ξεκινήσουν διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό θα καταστεί δυνατόν να συμμετέχουν στην έλυση αξία. Και φυσικά χρειαζόμαστε μια ευρύτερη πρόπτικη και όχι ένα περιορισμό και μια αμφαλοσκόπηση στα ευρωπαϊκά ζητήματα, γιατί είμαστε τμήμα μιας παγκόσμιας αγοράς. Και όντως η στρατηγική αυτή, η ευρωπαϊκή στρατηγική έχει μια παγκόσμια σκοπιά για το εμπόριο και υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για να εξασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού και δίκαιος ανταγωνισμός. Υπάρχουν ενδιαφέροντα μέτρα όπως η εξέταση των, ε, των εξωτερικών επενδύσεων, των ξένων μάλλον επενδύσεων και υπάρχει μία μάχη προάσπισης των ευρωπαϊκών αξιών και ελπίζω να στεφθεί με επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Το εκτιμούμε και πιστεύω ότι θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας και άλλες μελέτες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την παρουσίαση. Well, the uh, Το επόμενο θέμα αφορά την παρουσίαση της μελέτης ε, του προγράμματος Γαλιλαίου από τη ΣΤΟΑ. Ο of the Ο δόκτωρ μηχανικός Ουλφ Μπέστμαν ε, θα μας παρουσιάσει τη μελέτη. Σας ευχαριστούμε που Ήρθατε, εργάζεται στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Braunschweig, ε, στο Ινστιτούτο Κατεύθυνση Τροχιά από το 2003 και είναι επικεφαλή τη ομάδα πλοήγηση και αναπληρωτή διευθυντή ε, ε, του Ινστιτούτου. Εργάζεται στην πλοήγηση με δορυφόρους σε συστήματα μέτρησης σε πραγματικό χρόνο και είναι εξειδικευμένο στον τομέα της πλοήγησης. Η σημερινή μελέτη προετοιμάστηκε για τη ΣΤΟΕ το 2018 προκειμένου να δώσει το απαραίτητο ιστορικό για να κατανοήσουμε τις αρχές εργασίας του GNSS, του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης και για να τονιστούν οι ιδιότητες του Γαλιλαίου σε σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Η μελέτη είναι σχετική με την εργασία της Επιτροπής μας καθώς προετοιμάζουμε την ακρόαση της υποψήφια επιτρόπου για την ιστορική αγορά με ένα σημαντικό ρόλο για το διάστημα στο χαρτοφυλακιό τη και επίσης θα ολοκληρώσουμε και τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Χωρίς χρονοτριβή, έχετε το λόγο κύριε Μπέστημαν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή μου να απευθύνομαι εδώ σήμερα σε εσά για τη μελέτη μας για το ε, Γαλιλαίο και την ε, ε, επιστροφή της επενδύσεις για τις εφαρμογές στο διάστημα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η ημερήσια διαταξή μου έχει την εξή δομή. Καταρχήν θα σα κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το Γαλιλαίο και για άλλα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης παγκόσμια ε, κατόπιν ε, εξετάζουμε ε, τις εφαρμογές του Γαλιλαίου σε διάφορους τομείς και θα σας παρουσιάσω τις διάφορες απαιτήσει των διαφορών τομέων. Κατόπιν θα σας παρουσιάσω τα ωφέλη που μπορεί να έχει το Γαλιλαίο αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα και βάσει αυτού θα παρουσιάσουμε 7 στόχους πολιτικής και απόψεις τα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, το GNSS, είναι μια τεχνολογία κλειδί για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τη διασφάλιση της βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Επιτρέπει στους χρήστες του GNSS να καθορίσουν τη θέση τους παγκοσμίω. Ε, αποτελεί ένα δομικό μπλοκ της σημερινής υποδομής το Γαλιλαίο και τα συστατικά συστήματα αποτελείται από δορυφόρους ε, σε τροχιάς ε, που ε, στέλνουν διάφορα σήματα. Μπορούν οι χρήστες να βρουν τη δική τους θέση και επίσης λαμβάνουν και μηνύματα. Σήμερα έχουμε τέσσερα ε, υφιστάμενα συστήματα, το Γαλιλαίο για την Ευρώπη, το GPS από τις Ηνωμένε Πολιτείε, το GLONASS από τη Ρωσία και το Μεντέν από την Κίνα. Ακόμη και αν όλα τα συστήματα έχουν ε, υψηλό επίπεδο συνεκτικότητας και διαλειτουργικότητας, υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές το Γκαλιλαίο ως ε, το Ευρωπαϊκό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Επιλογής έχει μοναδικά χαρακτηριστικά ε, σε σύγκριση με τα άλλα συστήματα. Έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί υπό με στρατιωτικό έλεγχο, ενώ όλα τα άλλα GNSS έχουν αναπτυχθεί ε, υπό στρατιωτική εποπτεία. Το Γαλιλαίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ε, μη στρατιωτικούς χρήστες ε, και είναι ε, η μόνη συστοιχεία GNSS που παρέχει τις υπηρεσίες σε μη στρατιωτικούς χρήστες και ε, ε, οι χειριστές του GPS και του Galileo έχουν ε, συμφωνήσει στο να υπάρχει ένα κοινό σήμα για το μέλλον. Ενώ το GPS βασίζεται μόνο στην μελλοντική γενιά δορυφόρων, το Galileo από την αρχή θα το χρησιμοποιήσει σε όλους τους δορυφόρους του. Το Γαλιλαίο, καθώς είναι μη στρατιωτικό σύστημα, ε, δίνει περισσότερες λεπτομέρειες ε, για την ε, αρχιτεκτονική και τα από ό,τι άλλα συστήματα. Αυτό βοηθά ιδίω για εφαρμογές υψηλής αποδοτικότητας υψηλής επιδόσεως ε, και ε, το Γαλιλαίο επίσης ε, όπως και το σύστημα Ζάζαρτ έχει υπηρεσία έρευνας και διάσωσης. Αυτή η υπηρεσία μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τα σήματα κινδύνου με ένα γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο. Όσο ποτέ στο παρελθόν. Επίσης, η υποδομή του Γαλιλαίου έχει μία μοναδική ικανότητα απάντηση έτσι ώστε οι χρήστε που είναι σε κίνδυνο να μπορούν να λάβουν μία απάντηση. Και προκειμένου να υπάρξει καλύτερη ασφάλεια, το το στοχεύει να εισαγάγει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας ε, για να διασφαλίσει ότι μπορούμε να ερευνήσουμε ε, κάποια σήματα. Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται σε εννέα τομείς εφαρμογής ε, του Γαλιλαίου. Έχουμε πάρει συνεντεύξεις από τους ειδικούς σε όλους τους συγκεκριμένους τομείς. Προκειμένου να κρατήσουμε ξεχωριστά τους διάφορους τομείς, έχουμε καθορίσει ένα σύνολο ε, δικτών βασικών επιδόσεων ε, ζητήθηκε από οι δείκτες ε, αυτοί ε, να καταστούν σημαντική από μη σημαντική και βλέπετε τα αποτελέσματα πάνω δεξιά στο διάγραμμα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι οι απαιτήσει διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τομέα και ανάλογα με την εφαρμογή. Έρχομαι τώρα στα ωφέλη του Γαλιλαίου για τους Ευρωπαίους πολίτες καθώς ε, είναι το μόνο δορυφορικό σύστημα προήγησης δορυφόρων υπό μη στρατιωτική διακυβέρνηση, προσφέρει κάποια ωφέλη που δεν μπορούν να προσφέρουν τα άλλα συστήματα. Παραδείγματο χάρη, έχουμε ακριβείς ε, πληροφορίες ε, που δεν είναι διαθέσιμες από άλλα GNSS. Αυτό βοηθά πάρα πολύ για κάποιες συγκεκριμένε εφαρμογές άλλα συστήματα μπορεί ε, εν μέρη να υποβαθμιστούν αν υπάρχουν πολιτικές εντάσεις, ε, παραδείγματος χάρη, ε, αν έχουμε προβλήματα για κρίσιμες ε, σε σχέση με την ασφάλεια ε, υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε σύγκριση με άλλα συστήματα πλοήγησης, δορυφορικά συστήματα, το Γαλιλαίο μπορεί να δώσει ε, αυξημένη ασφάλεια και βελτιωμένη ακρίβεια το Γαλιλαίο ε, αποτελεί την ευρωπαϊκή συνεισφορά στην, ε, στα διεθνή συστήματα παρακολούθησης κινδύνου. Ως ένα μοναδικό χαρακτηριστικό περιλαμβάνει και ένα back channel προκειμένου να ενημερώσει ένα άλλο διάβλο, δηλαδή για να ενημερώσει τους χρήστες ότι έχει λάβει το μήνυμά τους. Το λέω μπορεί να δοθεί ως ότι έχει κοινωνικονομικά ωφέλη, κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη σε διάφορα επίπεδα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Παρόλα τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη του Γαλιλαίου, υπάρχουν και κάποιες ε, προκλήσεις που παραμένουν από την τεχνική σκοπιά. Το Γαλιλαίο όπως ε, κάθε άλλο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, είναι ιδιαίτερα ευπαθές σε παρεμβολές ραδιοσυχνότητας. RFI λέγονται. Αυτό σημαίνει ότι πολύ απλές ε, συσκευές μπορούν να διακόψουν τις υπηρεσίες ε, σε ένα ευρύ επίπεδο. Επίσης, απαιτεί πιστοποίηση των καλλιών για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη οι εφαρμογές για την αεροπλοεία Γι' αυτό η ενηχνευσιμότητα όλων των συνιστοσών και των απαιτήσεων είναι ε, σημαντική, αλλά δεν εφαρμόζεται πλήρως ακόμη. Σε ό,τι αφορά τώρα την επικοινωνία. Τα έγγραφα αναφορά στο Γαλιλαίο αποτελούν ε, έγγραφα ελέγχου της διαπαφής και έγγραφα που αφορούν τις επιδόσεις. Ε, Κάποιες ε, λεπτομέρειες όμως που είναι απαραίτητες για κάποιες εφαρμογές δεν ε, έχουν συμπεριληφθεί ακόμη στο έγγραφο αυτό. Επιπρόσθετα, η διεθνής εναρμόνιση εμποδίζεται εν μέρη από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έγγραφα αυτά, στα έγγραφα αυτά. Επίσης, το Γαλιλαίο παρέχει εξαιρετική διαδικασία επικοινωνίας για να ενημερώσει τους χρήστες για τη σημερινή τους καθεστώς και τις αλλαγές. Παρ' όλα αυτά ε, δεν ε, αντικατοπτρίζονταν στην έκθεση αυτή όλα τα περιστατικά του παρελθόντος. Κάποιοι εμπειρογνώμονες είχαν ε, εκφράσει αμφιβολίες ότι φορά την οριμότητα αυτής της υποδομής. Αυτό συνδέεται άμεσα με κάποιες οργανωτικές προκλήσεις. Κάποιοι εμπειρογνώμονες παραπονούνται ότι οι χειριστές του Γαλιλαίου θα πρέπει να είναι πιο διαφανείς στο να επικοινωνούν ε, διάφορες δυσλειτουργίες του συστήματος. Παραδείγματο χάρη ε, για διάφορες ε, εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουμε τις ονομαστικές επιδόσεις του συστήματος πλοήγησης αλλά και τη συμπεριφορά του συστήματος σε περίπτωση που δεν λειτουργεί. Το Γαλιλαίο εξακολουθούσε να επέφερε στο παρελθόν από διάφορε αισιόδοξε προβλέψει υλοποίησή του. Ε, είχαμε αρχικού οδικού χάρτε πολύ φιλόδοξου που οδήγησε σε απώλειε σε διάφορα στάδια και τώρα αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Επομένω, ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για το μέλλον είναι κάτι απαραίτητο. Ερχόμαστε τώρα στους στόχους πολιτικής. Ο πρώτος στόχος πολιτικής αφορά την ελκυστικότητα του Γαλιλαίου. Όπως σας είπα, εξακολουθεί να υποφέρει σημαντικά το Γαλιλαίο από καθυστερήσεις σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να αντισταθμίσει τις καθυστερήσεις αυτές παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ελκυστικότητα για τους μελλοντικού χρήστες για να υπάρχει ευρύτερο ρόλο του Γαλιλαίου, κυρίως σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά συστήματα. Οι ενδυνάμοι χρήστε πρέπει να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα του Γαλιλαίου. Αυτό απαιτεί περαιτέρω προσπάθειες για να, να προωθηθούν οι αναπτύξεις του Γαλιλαίου για τους χρήστες σε διαφορούς τομείς επιπρόσθετα είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το Γαλιλαίο μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιείται από όλα τα είδη των χρηστών στο μέλλον. Και ιδιαίτερα σήμερα όταν ε, ανταγωνίζεται με άλλες ε, συστοιχίε GNSS ε, που είναι διαθέσιμες και σε χρήση. Το Γαλιλαίο επίσης θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει λεπτομερεί και ανοιχτέ πληροφορίε στους χρήστε επιπρόσθετα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και λεπτομερή χρονοδιαγράμματα είναι σημαντικά για όλους τους χρήστες ε, προκειμένου να μπορούν να σχεδιάσουν ε, την ένταξη των υπηρεσιών του Γαλιλαίου στα δικά τους προϊόντα και να αυξήσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης στο σύστημα Γαλιλαίο. Οι πολιτικοί θα πρέπει να διασφαλίσουν αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα για το Γαλιλαίο ακόμη και αφού το Γαλιλαίο θα έχει καταστεί πλήρως επιχειρησιακό. Στόχος πολιτικής 2. Η επαλήθευση σήματος είναι μοναδικό χαρακτηριστικό του Γαλιλαίου. Θέλει να διασφαλίσει ε, ότι υπάρχει ασφάλεια ε, και αποτρέπει κάποια ε, πλαστά σήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για διάφορες κρίσιμες εφαρμογές του Γαλιλαίου. Η σημερινή ανοιχτή υπηρεσία δεν παρέχει ακόμη επαλήθευση, ακόμη και αν έχει σχεδιαστεί να εφαρμοστεί αυτό στο εγγύς μέλλον προκειμένου να ε, μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας ε, θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω πρόωθηση. Επίσης, διάφορες μορφές επαλήθευσης ε, είναι δυνατές. Ε, το Γαλιλαίο είναι το μόνο GNS σήμερα που υποστηρίζει την επαλήθευση και την ε, ανάπτυξη χαρακτηριστικών ασφαλείας θα πρέπει να δοθεί έμφαση προκειμένου να διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτόν τον τομέα σε σύγκριση με τα άλλα δορυφορικά συστήματα. Τώρα έχουμε την ε, κυβερνητική υπηρεσία του Γαλιλαίου, το οποίο, ε, η οποία παρέχει αυξημένη ασφάλεια σε σχέση με τους υπόλοιπους. Όμως δεν ε, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα ποσοστά κρίσιμων υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επωφεληθούμε από τα ωφέλη αυτή τη υπηρεσία. Δηλαδή, θα πρέπει οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει να έχουν εύκολη πρόσβαση στην ανάπτυξη τη κυβερνητική υπηρεσία για κρίσιμε υποδομέ ή για άλλε συγκεκριμένε χρήσει. Αυτό θα συμπεριλάμβανε ε, το ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα έπαιρναν διαπίστευση PRS, κυβερνητικής υπηρεσίας και πρόσβαση στι σχετικέ πληροφορίες PRS. Περνάμε στο στόχο 4. Νέα χαρακτηριστικά του Γαλιλαίου. Τα νέα χαρακτηριστικά απαιτούν πρόσθετη προσπάθεια προκειμένου να αναπτυχθούν ε, νέοι ε, λήπτες, ε, προκειμένου να έχουμε ένα μια κατάλληλη λογία κόστους ανάλυσης. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι προσπάθειες και να προσθεθούν νέα χαρακτηριστικά στα σήματα Γαλιλαίου και στις λειτουργικότητες. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι να εφαρμοστούν ε, μελλοντικές υπηρεσίες υψηλής επιδόσης ε, όχι μόνο ε, σε μόνη ραδιοσυχνότητα αλλά σε πολλαπλές συχνότητες. Θα πρέπει να υπάρχουν λύτες. Έτσι λοιπόν η ανταγωνιστικότητα του Γαλιλαίου θα πρέπει να αυξηθεί παρέχοντας θέσεις, υπηρεσίες γεωντοπισμού για μεγάλο αριθμό χρηστών. Περνάμε στον στόχο 5 ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα επιλογήσης ε, που ε, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο ε, και έχουμε πολύ χαμηλή ισχύ του σήματος. Θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια απόλυτη απώλεια του σήματος θέσης για πολλούς χρήστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κατάλληλες λύσεις. Προτείνεται λοιπόν να υπάρχει ευαισθητοποίηση για τις λήψεις του GNSS γενικώ και να διερευνηθούν ε, βιώσιμες εφεδρικές στρατηγικές. Ε, ε, αυτά τα ανεξάρτητα συστήματα θα μπορούσαν να έχουν μετριασμένες αρνητικές επιπτώσεις αρνητικές πτυχές. Περνάμε τώρα στην πολιτική, στο στόχο πολιτικής 6. Έχουμε μικρές προσωπικές συσκευές ιδιωτικότητας και μέσα αν και η χρήση αυτών των συσκευών είναι παράνομη, χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερα στην πράξη επειδή είναι διαθέσιμες και επειδή υπάρχει ζήτηση από συγκεκριμένε ομάδες χρηστών. Προκειμένου ε, να καταπολεμήσουμε τα αποτελέσματα αυτών των συσκευών θα μπορούσαμε να έχουμε δύο στρατηγικέ Καταρχήν, να υπάρξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίχνευση και τον εντυπισμό αυτών των συσκευών. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε ένα ε, δίκτυο ε, συσκευών έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν αυτέ οι συσκευές, οι προσωπικέ συσκευές ιδιωτικότητα, PPDs. Επιπρόσθετα, οι συσκευές ιδιωτικότητα χρησιμοποιούνται ε, από διάφορα εταιρικά αυτοκίνητα για να αποφευχθεί η ανείχνευση θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ελκυστικότητα αυτών, της χρήσης αυτών των συσκευών. Και έρχομαι στην τελευταία διαφάνεια, στο στόχο πολιτικής 7 για εφαρμογές που είναι κρίσιμες για την ασφάλεια, κάποιες, απαιτούνται κάποιες διαδικασίες έγκρισης και επιστοποίησης. Έχουμε κατευθυντήριες γραβές, γραμμές πιστοποίησης ε, και διαδικασίες. Δεν είναι όμως δυνατό να χρησιμοποιηθεί το Γαλιλαίο στις εφαρμογές αυτές. Προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, το Γαλιλαίο θα πρέπει να ε, δώσει περισσότερες ε, πληροφορίες για τις επιδόσεις και για περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσλειτουργία. αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου μακροπρόθεσμοι, στους μακροπρόθεσμους κύκλους καινοτομίας σε τομείς όπως η αεροπλοεία, παραδείγματος χάρη γιατί μπορεί να χρειαστούμε μέχρι και 20 χρόνια μέχρι να ενταχθεί εντελώς η τεχνολογία αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμος να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Okay, thank you very much for your presentation. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση. Ε, θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις και μετά θα απαντήσετε. Η ναι, κυρία Καρβάγια. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σας. Έχω να κάνω μια γενική ερώτηση. Δύο χαρακτηριστικά του έργου αυτού είναι με, κοινά με άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα που περιλαμβάνουν πολλούς συμμετέχοντες και πολλές χώρες. Δηλαδή, Ε, η έλλειψη προγραμματισμού επίσης ότι χρειάζονται πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί και το άλλο είναι η έλλειψη ορατότητας δηλαδή αυτά είναι πολύ καλά για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αλλά δεν φαίνονται προς τα έξω στα κράτη-μέλη. Οπότε αν μπορέσετε να απαντήσετε σε αυτά τα τρία ερωτήματα θα σας ήμουν ευγνώμων για να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε στα μελλοντικά μεγάλα έργα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλή. Σας ευχαριστώ για την ε, παρατήρηση αυτή. για τα δεδομένα αυτά. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς μπορεί η νομοθεσία να βελτιώσει το Γαλλία να βελτιωθεί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μέσω της ερευνάς σας εάν είδατε ε, το τι συνέβη τον Ιούλιο του 2019 όπου είχαμε κάποια αποτυχία μέρους του συστήματος. Αν μπορούσαμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, αν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο και αν μάθαμε κάτι από αυτό, αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος ε, κίνδυνος για τα δεδομένα που ε, συλλέγονται εκεί για τους πολίτες ε, και τους ε, επιστήμονες ε, και βεβαίως αν υπάρχει κάποια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να αντιληφθούν και οι πολίτες το τι συμβαίνει και με το σύστημα ειδοποιήσεων το οποίο ενεργοποίησαμε μόλις στην Ελλάδα που ειδοποιούμε αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο ορατός πολίτες λέει η κυρία Καϊλή Ευχαριστώ ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν θέλετε. Κύριος κρούτλερ; Σας ευχαριστώ για τη μελέτη. Ε, είναι πολύ ανησυχητικό το συμπέρασμα της μελέτης σας. Φαίνεται υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων αρχών. Επίσης υπάρχει μια απώλεια εμπιστοσύνη των χρηστών. Βέβαια, όντω η καινοτομία φοβίζει πολλές φορές, το καινούριο φοβίζει. Αλλά το Γαλιλαίο θα πρέπει να δώσει μια πραγματική εναλλακτική λύση για το, σε σχέση με το GPS και να μην είναι συμπλήρωμα. Ε, και αν ε, επενδύσαμε 16 δισεκατομμύρια στο Γαλιλαίο, είναι για να είναι μια γνήσια και ανεξάρτητη λύση στο ε, GPS και όχι ένα συμπλήρωμα του GPS. Επίσης, ότι είναι είπατε ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση της διακυβέρνηση και σίγουρα και το απόγευμα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Είχαμε φυσικά τη βλάβη του Ιουλίου, αλλά και αρχές Σεπτεμβρίου είχαμε ένα άλλο πρόβλημα που ανέκυψε. Οπότε διακυβέρνηση, σημαντικό θέμα, ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών από τις υποδομές που έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσε οι συστάσεις σας στο τέλος. Σίγουρα πολλά θα πρέπει να γίνουν ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να χρησιμοποιούν το Γαλιλαίο θα πρέπει να είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και... Το κύριο Στουσανόφσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση αυτή που μας κάνατε. Χαίρομαι ιδιαίτερως για την μελέτη αυτή και για το ότι την παρουσιάζετε στην Ήτρα γιατί ήμουν και στο πάνελ της ΣΤΟΑ, ε, είχα ξεκινήσει την έκθεση αυτή, ε, την οποία τη δέχτηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι συνάδελφοι. Είναι λοιπόν μια σημαντική αυτή η μελέτη. Ε, λόγω ακριβώς αυτού του στοιχείου της κριτικής που ασκείται δηλαδή στα πράγματα που περιπλέκουν τον Γαλιλαίο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα ξεκινήσει εύκολα γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα ακόμα. μέσω τον Γαλιλαίο έχει γίνει τμήμα των δημόσιων υποδομών. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη που αρχικά δεν είχε προγραμματιστεί. Πριν από πολλά χρόνια ήμουν εισηγητής ε, για το Γαλιλαίο και τότε ο στόχος ήταν να είναι ένα εμπορικό έργο. Και είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες με αυτό. Οπότε είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένος που ε, έχει πλέον ε, χαρακτηριστεί ως ένα έργο δημόσιων υποδομών. Τα όλα αυτά, εντάξει, είναι κάτι το οποίο αφορά το μέλλον και δεν μπορούμε να συλλάβουμε ακόμα τις εφαρμογές που θα έχει. Έχουμε λοιπόν και τις επιτυχίες και τα προβλήματα του Γαλιλαίου. Οπότε η ερώτησή μου είναι ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιλογές για συνεργασία με άλλα έργα όπως τον Κοπέρνικο και άλλα έργα υποδομών. Νομίζω ότι μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε τα διάφορα ωφέλη που θα έχουμε μπορούμε να, θα μπορέσουν να εμφανιστούν νέα προϊόντα. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας έχοντας κάνει αυτή την μελέτη για την περαιτέρω ανάπτυξη του καλλιλίου και της χρήση του μας με τα άλλα ευρωπαϊκά συστήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Κασάρης. Γεια σας. Ευχαριστώ θερμά για την μελέτη ευρυθής ε, μελέτη. Μας παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά του Γαλιλαίου και τα ωφέλη του στις μεταφορές, στην ασφάλεια, στον πολιτισμό, στη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε αμέριστα και εξακολουθεί να στηρίζει το Γαλιλαίο. Βέβαια, εντοπίσατε μια σειρά προκλήσεων και τις ε, είδαμε και εμείς ε, αυτές τις προκλήσεις. Όπως είπε και η συνάδελφος Εύα Καϊλή, το, τον, τον Ιούλιο είχαμε ένα συμβάν ε, και περιμένουμε ακόμη τα συμπεράσματα αν έγινε κάποια αντλήση διδαγμάτων από το επεισόδιο αυτό και επίσης η συμβολή του στην ανάπτυξη κάποιων βασικών εφαρμόγων. Εμείς θα θέλαμε να γίνει σημείο αναφοράς το Γαλιλαίο και με τα προβλήματα που αντιμετώπισε, διαπιστώσαμε ότι για να γίνει σημείο αναφορά στο Γαλιλαίο θα πρέπει να σημειώσει περισσότερη πρόοδο και να γίνει απόλυτα λειτουργικό. Γιατί είδαμε ότι φέτο ε, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα τμήμα και το 2021 θα ολοκληρωθεί. Αυτή η καθυστέρηση δεν είναι θετική, γιατί όχι μόνο πραγματοποίησαμε γενναιόδορες επενδύσεις, αλλά περιμέναμε και κάποια απόσβευση, κάποιο όφελος και προς το παρόν δεν βλέπουμε τέτοια αξιοποίηση των επενδύσεων. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχουν προβλήματα κυβερνοασφάλειας. Με τις προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας, πιστεύετε θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον ΕΝΙΣΑ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας. Και τέλος, είχαμε και πρόσφατα ένα συμβάν. Ε, πριν λίγες μέρες, ε, στη Σαουδική Αραβία, ε, επίθεση κατά των δηληστηρίων πετρελαίου. Είναι δυνατόν λοιπόν να ελέγξουμε drones που χρησιμοποιούνται για τις επιθέσεις ε, μη στρατιωτικών στόχων ε, μέσω της χρήσης του Γαλιλαίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος άλλος? Αν όχι. Κύριε καθηγητά. Ε. Παρακαλώ απαντήστε. Ναι, ναι. Πολλές ε, και διαφορετικές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τον προϋπολογισμό. Κατά την άποψή μου έχει μεγάλη σημασία να συνεχιστεί η προσπάθεια και η χρηματοδότηση του Γαλιλαίου γιατί έχουμε επενδύσει ήδη πολλά λεφτά αλλά ήδη βλέπουμε πως υπάρχει μια αγορά λιανικής και βγάζουμε πολύ περισσότερα λεφτά με τις νέες αυτές ε, τεχνολογίες. και αυτό μας δίνει ένα όφελος ε, και εσόδων από την πνευματική ιδιοκτησία για τα ευρωπαϊκά κράτη και την ευρωπαϊκή βιομηχανία για το μέλλον. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε ε, βασική περιοχή του κόσμου στον τομέα της έρευνας για προϊόντα δορυφορικής πλοήγησης όπως με ενημερώνουν. Οπότε τώρα θα μιλήσω γερμανικά, μου επιτρέπετε. Η επόμενη ερώτηση αφορά το θέμα της ορατότητας ε, του Γαλιλαίου. Οπωσδήποτε αυτό είναι ένα πρόβλημα με την έννοια ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει να έχει μια εφαρμογή στο κινητό ε, και είναι ήδη με GPS και δεν ε, παρακολουθεί καμία, δεν βλέπει καμία διαφορά ε, αν το κινητό κάνει την ε, πλοήγηση με το Γαλιλαίο και δεν θα είναι άμεσα και ορατές η... Ε, δεν θα είναι άμεσα ορατά τα πλέον εκτίματα στον τομέα της ακρίβειας αν μιλάμε για το κινητό συγκεκριμένα. Οπότε το θέμα είναι ποιες επιπλέον εγγύησης ασφαλείας ε, και πολιτικά πλεονεκτήματα παρέχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Γαλλίο γιατί έχουμε αρκετές κρίσιμες υποδομές σήμερα οι οποίες εξαρτώνται από την χρήση δορυφορικής ε, πλοήγησης να σκεφτούμε τον συγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρισμού, των δικτύων ε, κίνητης τηλεφωνίας όλα αυτά σήμερα βασίζονται σε σήματα της δορυφορικής ε, πλοήγησης που αφορούν ε, τον ακριβή χρονισμό ή προσγείωση των αεροπλανών επίσης. Ε, εδώ πέρα λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Γαλλίο και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας επίσης και σε άλλους. Πρέπει λοιπόν να αναλυφθούν περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε να αντιληφθεί ο Ευρωπαίος πολίτης πως όλες αυτές οι τεχνολογίες βασίζονται στην ε, δορυφορική πλοήγηση και μακροπρόθεσμα το Γαλλαίο ε, προσφέρει ένα πλεονέκτημα γιατί τα συστήματα αυτά δεν μπορούν έτσι απλά να αφαιρεθούν ε, και ο πολίτης θέλει να έχει το σύστημα στο χέρι του οπωσδήποτε. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στις διάφορες ερωτήσεις ε, που αφορούν ε, την πτώση του συστήματος ε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Βεβαίως, ως επιστήμονας του Πανεπιστημίου Μπανασφάκη δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς στην ΕΖΑ. Ανεξαρτήτως αυτού βεβαίως βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τι επιδράσεις είχε ε, το ότι έπεσε το σύστημα. Αν δούμε, παραδείγματος χάρη, τον δικό μου τον τομέα της αεροπορίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν η διακοπή η ίδια γιατί συστήματα που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια ε, πρέπει να μπορούν να συνεχίζουν τη λειτουργία τους ε, ακόμα και αν διακοπεί η λειτουργία ενός μέρους του συστήματος πολύ πιο δραματικό σε τελική ανάλυση ήταν το θέμα της επικοινωνίας ε, κατά τη διάρκεια της ακοπής λειτουργίας. Δεν υπήρξε κάποια προειδοποίηση ούτε από το σύστημα, ούτε κανονικά αυτό γίνεται εντός ε, των συστημάτων ε, που λαμβάνουν τα σήματα των δορυφόρων και ελέγχουν την υγεία του συστήματος ε, και δεν λειτουργήσαν. Βεβαίως αυτό είναι πρόβλημα γιατί πλέον ε, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στους δείκτες αυτούς. Επιπλέον ε, υπάρχουν ήδη κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας που θα πρέπει να μεταδίδουν ακριβώς τέτοιες τις λειτουργίες τους χρήστες. Ε, διάβλοι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ αργά και όχι αρκετά. Δηλαδή, κανονικά θα ανέμενε κανείς ε, πριν φτάσουμε σε μια τέτοια κρίσιμη διαταραχή να έχουμε μια ειδοποίηση στους ε, χρήστες ε, είναι κάτι το σύνηθες στην αεροπορία ε, πριν την άφηξη ξέρω εγώ μιας πτήσης όπως γίνεται παραδείγματος χάρη και πριν από το ταξίδι ενός αυτοματοποιημένου αυτοκινήτου να υπάρχει μία ειδοποίηση και να γίνεται χρήση μόνο όταν είναι λειτουργικό το σύστημα και αναλόγως ε, λοιπόν θα πρέπει τα συστήματα αυτά πληροφόρησης να λειτουργήσουν καλύτερα και να δίνονται περισσότερες ε, λεπτομέρειες για την κατάσταση του συστήματος και την διάρκεια της διακοπής ε, λειτουργίας. Αυτό είναι περισσότερο το πρόβλημα. Η διακοπή η ίδια, εντάξει, μπορεί να συμβεί και ακόμα και σε συστήματα κρίσιμα για την ε, ασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται. Ένα άλλο ερώτημα ε, πάει προς την κατεύθυνση του ποιο πλεονέκτημα έχει το Γαλιλαίο απέναντι στο GPS. Έχουμε ήδη πάρα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορεί να μας προσφέρει αν υπάρχουν ας δυνατότητες ε, στο GPS να επιδεινωθεί το σήμα η λεγόμενη επιλεκτική διαθεσιμότητα. Ε, υπάρχουν ίσως σήμερα άλλες δυνατότητες για να επηρεαστεί το σήμα. παραδείγματος χάρη σε περιοχές στις οποίες λαμβάνουν χώρα στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το αρχικό σύστημα το είχε σβήσει ο Αμερικανικός στρατός ε, ως ε, απάντηση στην ενεργοποίηση του Γαλιλαίου κατόπιν εντολής του Προέδρου Κλίντον. Δηλαδή, αν ε, δεν υπήρχε το Γαλιλαίο θα ε, υπήρχε σήμερα αυτή η επιδείνωση γιατί δεν υπήρχε κάποιος λόγος για να κλείσει το παλαιότερο σύστημα Απλά ήθελαν οι να εμποδίσουν την εξέλιξη του Γαλιλαίου. Και εδώ πέρα βλέπετε λοιπόν ποια στρατηγική αξία έχει ένα τέτοιο σύστημα για διάφορες χώρες. Επιπλέον, το Γαλιλαίο ήδη σήμερα έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν έχουν άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Παραδείγματος χάρη στο GPS και στο GLONASS ε, έχουμε μία συχνότητα την L1 που είναι αφιερωμένη στην αεροπορία. Το Γαλιλαίο μας προσφέρει στην αεροπορία πάντας, ε, πάντα μιλώντας περισσότερα σήματα στην συχνότητα L1 και L5. Τα σήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διορθωθούν ε, σφάλματα του σήματος και προσφέρουν ε, έτσι περισσότερες επιλογές γιατί οι δορυφόροι του Γαλιλαίου ευθύς εξ αρχής ε, είχαν αυτό το χαρακτηριστικό άμεση αντίδραση ε, δε σε αυτό ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχουν ε, ανάλογες δυνατότητες και σε μελλοντικούς δορυφόρους του GPS. Εδώ πέρα λοιπόν το Γαλιλαίο έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στο σύστημα GPS, ε, το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε δηλαδή στο σύστημα αυτό στο σύστημα το GPS οι νέες συχνότητες θα πρέπει να εφαρμοστούν με την εκτόξευση κάθε νέου δορυφόρου. Δηλαδή μιλάμε για μια δεκαετία ίσως για να φτάσουν όλοι οι δορυφόροι να εκπέμπουν στην συχνότητα L5. Οπότε ο Γαλιλαίο έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα απέναντι στο σύστημα GPS γιατί παρέχει αυτό το χαρακτηριστικό ήδη σήμερα στους ε, χρήστες και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να προωθήσουμε ακριβώς το σύστημα και να αυξήσουμε την ελκυστικότητα του συστήματος μας για τους ε, χρήστες. άλλη ερώτηση αφορά το σύστημα backup. Το Γαλιλαίο έχει κάποιες αδυναμίες που έχουν όλα τα συστήματα δορυφορικής ε, πλοήγησης, ε, δηλαδή μπορεί να υποστεί επίγειες παρεμβολές, ε, μπορεί να υποστεί παρεμβολές από τους ηλιακούς ανέμους που μπορεί να επηρεάσουν το σύστημα. Γι' αυτό Μία επιλογή πολιτικής ε, ήταν ε, πέρα από την ε, εξέλιξη του Γαλιλαίου μελλοντικά να δούμε και άλλες τεχνολογίες πλοήγησης που θα δώσουν ανεξάρτητες δυνατότητες εντοπισμού στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας ε, του συστήματος Γαλλίου ή όλων των ε, συστημάτων ε, δορυφορικής πλοήγησης παραδείγματος χάρη μια που τα συστήματα μετάδοση του ρεύματο βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό μια πάυση λειτουργίας θα είχε πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες επίσης στην αεροπορία αναμένουμε ανάλογες ε, συνέπειες ε, εάν ε, και εκεί τα επιπρόσθετα στήματα ναυτιλίας σταματήσουν να λειτουργούν. Οπότε, κατά την άποψή μας, το Γαλιλαίο ήδη σήμερα είναι μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δείξει ότι έχουμε και μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα πάρα πολύ αποδοτικό και η αντίδραση των άλλων διαχειριστών ε, παγκοσμίων ε, συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης μας δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Μια άλλη ερώτηση αφορούσε το θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας και της χρήσης του Γαλιλαίου για τρομοκρατικές επιθέσεις. σε σχέση με την ε, κυβερνοασφάλεια πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Αφενός ε, η χρήση του Γαλιλαίου, η κατάχρηση μάλλον, για σκοπούς ε, ανεπιθύμητους, όπως παραδείγματος χάρη το να κατευθύνει κάποιος drone σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οπωσδήποτε ένα τέτοιο ανοιχτό σύστημα ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους χρήστες. Και ένα σύστημα για αποφυγή τέτοιας κατάχρησης θα πρέπει να έχει μια άλλη μορφή. Αλλιώς ε, θα περιορίζαμε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα, ανεξαρτήτως του τι ίσως ε, είδατε ε, στην ε, Σαουδική Αραβία που ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει με ή χωρίς το Γαλιλαίο. Η άλλη πτυχή είναι η επίθεση στο ίδιο το σύστημα. Ανέφερα, είδα πως, ανέφερα ήδη πως έχουμε κρίσιμες υποδομές που εξαρτώνται από αυτήν την τεχνολογία υπάρχουν ε, διάφορες δυνατότητες παρέμβασης στο σύστημα από την απλή παρεμβολή του σήματος όπου πρέπει να αναπτύξουμε κάποιες στρατηγικές εναλλακτικές με ως ε, την ε, παραποίηση του σήματος σε αυτό το Γαλιλαίο είναι το μόνο σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει την δυνατότητα κρυπτογράφησης ε, και ταυτοποίησης του σήματος του. Είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προωθήσουμε την ε, χρήση του Γαλιλαίου. Εδώ πέρα λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχουν εγκαίρως περισσότερες πληροφορίες για τους δυνητικούς χρήστες Μιλάμε για μια σειρά εφαρμογών που μπορούν να έχουν οι χρήστες όπως παραδείγματο χάρη το να έχουν διάφορα συστήματα χρονικής σφραγίδα κάτι το οποίο είναι ήδη υποχρέωση στα χρηματοοικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ας πούμε. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Εμείς σας ευχαριστούμε, Δόκτωρα Μπέστμαν. Ευχαριστούμε και για την παρουσίαση της μελέτης και για τις διεξοδικές διευκρινήσεις. Σίγουρα θα συνεχιστεί η συζήτηση για το Γαλιλαίο, γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος και το θέμα αυτό και οι εφαρμογές του και όλα τα συναφή με το Διεθνές Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, διεκπαιρεώσαμε την πρωινή μας ημέρη σε διάταξη, αλλά και το απόγευμα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θα μιλήσουμε για το διάστημα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ραντεβού λοιπόν στις 2.30 και πάλι. Καλό σας μεσημέρι και καλή όρεξη.